ώστε να μην έχουμε τόσο θόρυβο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις της ψήφου. Θα ξεκινήσω σε 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε τώρα στις διολογήσεις ψήφου. Πρώτο θέμα είναι η σύσταση Βαλένσα για την Συμφωνία Σύμπραξη στον τομέα της βιώσιμης ελίας μεταξύ Ένωσης και της Λιβερίας. Για ένα λεπτό, ο κύριος Ζαν Λουκ Μελανσόν πρώτος. Σε Λοιπόν, αντιτίθεμαι σε αυτό το κείμενο, διότι έχουμε αυτή τη λογική παρέμβαση της Ευρώπης στους φυσικούς πόρους ορισμένων χωρών και στην περίπτωση της Λιβερίας η κατάσταση είναι ακόμη πιο απαράδεκτη. Το 50% του τοπικού πληθυσμού, ξέρετε, ζει από την αλία και εμείς επιτρέψαμε να αλλιεύονται 3.500 τόνοι τόνου που θα αφαιρεθούν από τους ε, ντόπιου και τους αφαιρούμε τις δυνατότητες να ζήσουν ε, όλο αυτό είναι κατά των τοπικών πληθυσμών Ευχαριστούμε Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Άντρες Μάμικινς για ένα λεπτό σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στον ε, Ευρωπαίο ψαρά να ψαρεύει νομίμως στην οικονομική ζώνη της Λιβερίας και θα βελτιώσει ταυτόχρονα την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών ειδικά όσον αφορά τον τόνο. Μάλιστα στην ε, Λιβερία 12% του ΑΕΠ παράγεται από την Αλία και είναι ένα πολύ μικρό ποσό και η Αλία θα μπορούσε να παίξει πολύ σοβαρότερο ρόλο στην οικονομία της Λιβερίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνιελ Χάναν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε ε, για το ότι θα πάμε να ψαρέψουμε τα ψάρια άλλων είναι λόγω της καταστροφής που έφερε η κοινή αλληλευτική πολιτική στα δικά μας ύδατα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την αλληλευτική πολιτική ως ένα σύμπτωμα ευρύτερων προβλημάτων. Δηλαδή το πώς προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις, ε, τους πρακτικούς περιορισμούς. Εξακολουθούμε λοιπόν να έχουμε αυτή τη μανία με την αρχή ενός κοινού πόρου στον οποίο όλοι έχουν πρόσβαση όπως ακριβώς διατηρούμε το ευρώ παρά την δυστυχία που φέρνει σε αυτούς που το χρησιμοποιούν, όπως διατηρούμε την Σέγγεν παρά τα προφανή μεταναστευτικά προβλήματα που δημιουργεί, γιατί τα πάντα θυσιάζονται στο δόγμα της ολοένα και στενότερης ένωσης. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε πως παρά τις προφανείς καταστροφές στη Βρετανική αλληλεία, η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν ήταν αντικείμενο της πρόσφατης διαπραγμάτευσης. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Σας ευχαριστώ. Στέφανο Μάουλο για ένα λεπτό. Α, μάλιστα. Ο κύριος Μάουλο δεν θα μιλήσει μου λένε. James Carver λοιπόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα βεβαίως, βεβαίως καταψήφισα Βλέπουμε την καταστροφή που υπάρχει, την οικονομική και την περιβαλλοντική της κοινή αλλιευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα κάνουμε και εξαγωγή στην Δυτική Αφρική. Και ακόμη παραπέρα βλέπουμε ότι έχουν κάνει αλληλευτικές συμφωνίες σε άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής. Δεν βοηθάμε έτσι τις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου. Ε, βλέπουμε 600.000 ευρώ που πάνε κάθε χρόνο σε 34 μόλις σκάφη για να αλλιεύσουν 600.000 τόνους ψαριών. Μα τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα στους ψαράδες της Λιβερίας. Φοβάμαι ότι θα έχει, ελπίζω δηλαδή να μην έχει τα ίδια αποτελέσματα που είχε σε πολλά άλλα μέρη της Δυτικής Αφρικής όπου όχι μόνο ψα... τα δικά τους αλλιεύματα αλλά τους σκοτώνουν τα ευρωπαϊκά ψαροκάικα. Είναι έσχος και ανθρωπιστική καταστροφή. Περνάμε τώρα στην επόμενη σύσταση του κυρίου Γκαμπριελ Μάτο. Συμφωνία ληφτικής σύμπραξης με την Μαυριτανία. Δύο είναι οι ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Μάμικιντς για ένα λεπτό. Ε, ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη συμφωνία συναφθήκε το 89. Ακολούθησαν ε, και άλλες συμφωνίες στη συνέχεια. Επιχειρήσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά δυστυχώς η Μαυριτανία Ε, καταφέρεται κατά της ε, εκφόρτωσης των Λασπάλμας ε, στα Καναρία Εμείς θεωρητικά καταλαβαίνουμε τη λογική μιας τέτοιας απόφασης, αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα στις επόμενες συνεδριάσεις επιτροπής. Επειδή η Μαυριτανία δεν κατέχει αναπτυγμένες υποδομές, όπως απαιτούνται. Αυτή η απέτηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης είναι παράλογη, αλλά εγώ είμαι υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντάνιελ Χάναν για ένα λεπτό. Δεν είναι πια στην αίθουσα μάλλον. Οπότε, περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Τόμασιτς. Νέα μέσα για την δαφική πολιτική συνοχής. Η κυρία Μόρβα έχει πρώτο λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επινοεί τακτικά τέτοιες έννοιες που υποτίθεται ότι είναι επαναστατικές πολιτικές και υπόσχονται αλλαγή. Αυτό έχω δει εγώ την τελευταία επτά Αλλά αυτό που έχω δει επίσης είναι ότι για το λαό τίποτα δεν βελτιώνεται. Σίγουρα όχι για του επωνομαζόμενου ε, δεύτερης κατηγορία πολίτε ε, στα επωνομαζόμενα δεύτερης κατηγορίας κρατήμελη. Εδώ μιλάμε για την πολιτική συνοχή, αυτή είναι η έννοια κλειδί και μιλάμε για τοπική ανάπτυξη και μιλάμε για την ε, CLLD, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Ωραία λόγια, αλλά αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι ότι βάζει εμπόδια στι χώρε αυτέ όπω την Ουγγαρία. Πώ μπορούμε να μιλάμε για τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, σε κοινότητε όπου έχει κλαπεί γη. Δεν υπάρχει πια ουγγρική γη. Όλη η γη ανήκει σε ξένου. Ούτε μικρομεσαίε επιχειρήσει υπάρχουν λόγω των πολυεθνικών ε, ομίλων που έχουν καταστρέψει τι μικρέ επιχειρήσει. Ούτε έχουμε καλού ηγέτε πια, διότι εκπαιδευμένοι άνθρωποι έχουν φύγει από τι χώρε του και πάνε να δουλέψουν αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος... για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε, στην, περίοδο, στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε μια ολοκληρωμένη δαφική προσέγγιση για την πολιτική συνοχής. Δύο είναι τα νέα μέσα, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, το CLLD και το ITI. Χρησιμοποιούνται στο υποπεριφερειακό επίπεδο ώστε να βοηθήσουν τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης αυτής της στρατηγικής ε, μέσω της χρήσης πόρων από διάφορες πηγές. Τώρα το 5% έχει δεσμευτεί, μιλάμε για 16 δις ευρώ και εγώ το υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μακοβέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η συνθήκη της Λισαβόνας του 2008 προβλέπει ότι η εδαφική συνοχή αποτελεί ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική συνοχής και από διαρθρωτικά ταμεία, από αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων για να μην έχουμε αποκλήσει στην ανάπτυξη των διαφόρων επικρατιών και περιφερειών και να έχουμε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στην περίοδο 2014-2020 έχουμε περισσότερα εργαλεία για ΣΔΙΤ, για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και για υφόρες επενδύσεις. Μπορούν λοιπόν να δημιουργήσουν δίκτυα οι πόλεις, οι νομοί, και έτσι να δουλέψουν προς την ανάπτυξη. Τα κράτη δίνουν προτεραιότητα στις συνδέσεις, στη συνδεσιμότητα με τον πυρήνα της Ευρώπης, σε βάρος των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε για περισσότερη εδαφική ολοκλήρωση. Στη Ρουμανία το 47% του πληθυσμού ζει στην Ήπεθρο και θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές για να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ντάνιελ Χάναν, δεν είναι στην αίθουσα. Λοιπόν, yes, υπόσπιση για ένα λεπτό. Δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο. Εδώ μιλάμε για τη, ε, ε, ε, ταμεία της διαρθρωτικής πολιτικής τα οποία δεν έχουν πάντα σωστά αποτελέσματα ούτε γίνονται με σωστών έργων. Είμαι βέβαιος όμως ότι η πολιτική αυτή έχει νόημα και ότι οι θετικές πτυχές θα κυριαρχήσουν στις αρνητικές. Γι' αυτό υποστήριξα αυτή την έκθεση και καλωσορίζω τα νέα εργαλεία που εισάγονται και που θα γίνουν διαθέσιμα για τους Δήμους μέσω των οποίων θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα χρηματοδότησης των έργων τους. Φυσικά το ποσοστό αποτελεσματικότητας θα πρέπει να το παρακολουθούμε διότι σίγουρα υπάρχουν ε, προγράμματα αμφίβολης ε, αποτελεσματικότητας Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος ε, για τις πόλεις και τους δήμους μας διότι μερικές φορές ε, για λόγους ε, γραφειοκρατίας δεν μπορούν να πάρουν τη χρηματοδότηση κάποιες πόλεις. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται πως και ο κύριος Μάουλο και ο κύριος Πόλτσακ δεν είναι πια στην αίθουσα. Πεινούσαν μάλλον. Εντάξει, τους το συγχωρώ. Ο κύριος Έφριτς λοιπόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταψήφισα τα μέτρα αυτά. Όπως καταψηφίζω οτιδήποτε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην οποία είμαι μέλος, για ένα πάρα πολύ απλό θέμα αρχής. Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου πληρώνει τους φόρους του και πρέπει να πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι να τα μοιράζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπούμε εάν υπάρχουν φτωχές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά λυπούμε αλλά δεν πρέπει να τις χρηματοδοτούμε με τα λεφτά του Βρετανού φορολογούμενου. Έχουμε και δικά μας προβλήματα. Στο Midlands, από όπου κατάγομαι. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο γιατρό, δεν έχει σχολεία, τα, τους πετάνε έξω από τις εργατικές κατοικίες και τα λεφτά του Βρετανού φορολογούμενου τα μοιράζουμε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά καλό θα ήταν να τα πληρώνετε από την τσέπη σας, όχι από τη δικιά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην τελευταία έκθεση της κυρίας Ηλιάνας Γιώτοβα, πολιτική συνοχή στις ορεινές περιοχές. Για την Γκουε, εξ ονόματος της ομάδας, η κυρία Σένερα Ροντρίγκης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι αρκετά αμφίσιμη αυτή η έκθεση, περιλαμβάνει θετικά στοιχεία για τις ορεινές περιοχές, αναγνωρίζει βέβαια την ανάγκη στήριξης των αγροτών σε αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς όμως η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία εξαιρετικά αρνητικά. Σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα είναι ε, δημόσιους πόρους και δημόσια υπηρεσία υψηλής ποιότητας. Ιδαλλιώς δεν θα μπορεί να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές. Χρειαζόμαστε καθηγητές, χρειαζόμαστε προσωπικό στα εθνικά συστήματα υγείας για να έχουμε ε, ε, εκπαίδευση και υγεία στην υπεθροστή περιφέρεια και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ορεινές περιοχές βλέπουν τον πληθυσμό τους να τις εγκαταλείπει σιγά σιγά και οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις το μόνο που κάνουν είναι να προσπορίζονται όλους τους πόρους στις ορεινές περιοχές. Και δεν θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε αυτά με το προπέτασμα καπνού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και γι' αυτό καταψήφισα αυτή την έκθεση. Η Κριστίνα Μόρφεντ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι όσοι ζουν σε φτωχές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένες περιοχές θα πρέπει να έρθουν κοντά με άλλους, θα πρέπει να βοηθηθούν και γι' αυτό χρειαζόμαστε σωστή στρατηγική. Θα έπρεπε ήδη να κάνουμε κάτι τέτοιο τα τελευταία δέκα χρόνια, όχι μόνο για τις ορεινές περιοχές, αλλά για όλες τις χώρες που υστερούν, που καθυστερούν, που τα επίπεδα ανάπτυξής τους δεν είναι τόσο υψηλά όσο θα έπρεπε. Και δεν υπήρχε υπάρξει καθόλου μείωση της απόκλησης μεταξύ αυτών των χωρών και των δυτικών χωρών της Ευρώπης και θα έπρεπε να έχει υπάρξει μείωση των αποκλήσεων αυτών. Να αναγνωρίσουμε πρώτα τις μειονεκτικές περιοχές, να τις εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά τυχαία. Δεν είναι ότι έχουν ενσκύψει φυσικές καταστροφές και έχει καταστραφεί η ύπεθρος. Καταστρέφεται η ύπεθρος γιατί υπάρχει αποπληθισμός, υπάρχει απερίμωση, την εγκαταλείμουν την ύπεθρο οι άνθρωποι λόγω της φιλελεύθερης, της νέο φιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελευθέρου εμπορίου χωρίς καμία προστασία των αδυνάμων. Κύριος Μάμικινς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ορεινές περιοχές είναι μόλις 30% της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά δυστυχώς δεν λαμβάνουν ειδική προσοχή αν δούμε την συνεισφορά τους στην οικονομία. Οπότε εγώ είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης. Θεωρώ πως θα πρέπει να αναπτύξουμε έναν ορισμό των ορεινών περιοχών στην πολιτική της συνοχής. Πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τις περιοχές αυτές όσον αφορά το πόσο αεροκατοικημένες είναι, να δούμε την ε, κλιματική αλλαγή και να δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν αν δούμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη για ένα λεπτό.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 Για αυτό το λόγο χρειάζεται μια νέα στρατηγική όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλιστεί η προστασία των περιοχών αυτών. συγχωρείτε, δεν υπάρχει διερμηνία σε κάποια γλώσσα. Περιμένετε λίγο. Δουλεύει τώρα. Ωραία. Κύριε Μακοβέη, μπορείτε να πάτε 30 δευτερόλεπτα πίσω και θα μηδενίσω το χρονόμετρο. Έχετε το λόγο. Μισό λεπτό ή ένα. Ξεκινήσω από την αρχή. Ε, χαίρομαι για αυτή την έκθεση διότι είναι προ όφελο τη Ρουμανία. Είναι προ όφελό μα να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι ορεινέ περιοχέ, στα Καρπάθια Όρη, στη Ρουμανία διότι χρειάζεται, χρειάζονται αυτές οι περιοχές ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ε, ώστε να αναπτυχθούν αλλά και για να προστατευτεί και το περιβάλλον των περιοχών αυτών. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποια στρατηγική για τις ορεινές περιοχές ούτε συνεπώς και για τα Καρπάθια. Θα ήθελα λοιπόν να εκπονηθεί μια τέτοια στρατηγική ώστε να υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια, σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις και να αναπτυχθούν οι ειρηνές μας περιοχές. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και την απασχόληση στις περιοχές αυτές. Ε, το συζητάμε διαρκώς, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ε, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη και επενδύσεις στις περιοχές αυτές. Περιοχές αυτές ε, που είναι πιο κατοικημένες βέβαια, αλλά που υπάρχει τουρισμός και ενδεχομένως και άλλες δραστηριότητες, άλλοι τομείς δραστηριότητας και άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ήταν η κυρά του Σιλίου Πόλτσακα, αλλά δεν είναι στην αίθουσα. Οπότε η Τελευταία είναι η Αντιπρόεδρος, η κυρία Μακίνεση, για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά εγώ ψήφισα υπέρ αυτή τη έκθεση διότι αφορά τη μέρημνα για τι απομακρυσμένε και ορεινές περιοχέ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω είπε μόλι η Μονικά Μονακοβέη, αυτό απαιτεί υπηρεσίε προ του κατοίκου των περιοχών αυτών, όπω ευρυζωνικέ υπηρεσίε, ιατρικέ υπηρεσίε, εκπαίδευση, υγεία, είναι λοιπόν πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή. Απασχόληση και ανεργία. Ανεργία, να υπάρχει υψηλό πρόβλημα ανεργία και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων στι περιοχέ αυτέ. Πώ θα διατηρήσουμε, κρατήσουμε και θα ενθαρρύνουμε του νέου να μείνουν σε αυτέ τι περιοχέ. Αν δεν έχουν δουλειέ, δεν θα μείνουν. Αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Και κάτι τελευταίο που σχετίζεται με την προηγούμενη συζήτηση για την ανεργία ε, πρέπει να εστιαστούμε ιδιαίτερα στους νέους στην Ιρλανδία. Έχουμε πρόβλημα διότι οι άνθρωποι με αναπηρίες αποκλείονται από το πρόγραμμα εγγύησης ε, για τους νέους. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης και ελπίζω οι υπουργοί μας να το ε, λάβουν υπόψη αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κανονικά δεν επιτρέπουμε χειροκροτήματα από τα θεωρία, αλλά μια που ήταν η τελευταία ομιλητή, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η συνεδρία θα επαναληφθεί στις 3. Καλή σας όρεξη.